την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ε, στην ε, υλοποίηση των συμπερασμάτων. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ε, συνάδελφοι, κλείνει η συζήτηση για τη Σρι Θα ψηφίσουμε μετά την συζήτηση και των υπόλοιπων ψηφισμάτων. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη το Αζερβαϊτζάν. Και δίνω το λόγο στην κυρία Βεζιά. Monsieur le Président, Κύριε Πρόεδρε, δεν συνηθίζω να μιλώ πρώτη και με έχει καταλάβει μια κάποια αμηχανία. Λοιπόν, για ε, πρώτη φορά, για μια ακόμη φορά μάλλον, συζητούμε την κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν. Η δημοκρατική κατάσταση στη χώρα αυτή είναι αρκετά δραματική. Είναι ωστόσο μια χώρα που είναι ένας μία μελιτέος εταίρος στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων της Ένωσης προς Ανατολάς η αντιπολίτευση, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει μιλούν για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και καταστολή, μιλούν για τη διαφθορά του καθεστώτο. Οι δημοκρατικέ αξίε, τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρητικά είναι αναπόσπαστο τμήμα των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπω λοιπόν θα έπρεπε να διδαχθούμε από αυτά που γίνονται στι λεγόμενε αραβικέ χώρε και να απαιτήσουμε από του ανατολικού μα εταίρου αυτό που δεν καταφέραμε να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση τη Τινησία, τη Λιβύης ή της Αιγύπτου. Μήπως κύριε Επίτροπε θα έπρεπε να φροντίσουμε η δημοκρατία τελικά να βασιλεύσει στις χώρες αυτές. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε κάποιες ελάχιστες απαιτήσει. ελάχιστε απαιτησει τωρα σε ό,τι αφορά το ψήφισμα, νομίζω ότι τουλάχιστον είναι, είναι ένα ψήφισμα των ελαχίστων. Δεν μας εκφράζει αυτό το ψήφισμα και γι' αυτό θα απόσχουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ, έχει λόγο. Κύριε Πρόεδρε, το Αζερβαϊτζάν δυστυχώς είναι ένα μονοκομματικό ή μη αυταρχικό κράτος και δεν γίνεται ανεκτή καμία κριτική. Οι περσινές εκλογές λογικά έδωσαν συντριπτική πλειοψηφία για το κόμμα του κυρίου Αλίγεφ. Ο ΑΣΕ είπε πως ε, δεν αποτελούν ουσιαστική πρόοδο εκλογές αυτές όσον αφορά τις δημοκρατικές εξελίξεις ήταν περιορισμένη η ελευθερία έκφρασης και οι φυσιολογικές πολιτικές συζητήσεις είναι αδύνατες λόγω των περιορισμών στον ΜΜΕ. Τώρα ακούμε, με συγχωρείτε κύριε Τάνοκ, λίγο πιο σιγά παρακαλώ για τις ερμηνείς. Ε, μα καταλαβαίνω αγγλικά εδώ μέσα ο κόσμος, λέει ο κύριος Τάνοκ. Ε, δεν μπορώ γιατί δεν θα μπορούσα να το διαβάσω όλο. Τώρα ακούμε τη στόχευση κομμάτων της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων. Απλά πρέπει που και που να θυμόμαστε εδώ πέρα τι είναι το καθεστώς αληγευ Είναι μια χώρα που όπως όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ανατολικής μας γειτονίας. Υποτίθεται λοιπόν πως έχει δεσμευτεί για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στην πραγματικότητα ξοδεύει πέτρο δολάρια για να πείσει τους ε, αλλοδαπούς για το πόσο καλό καθεστώς είναι. Εμένα δεν με ξεγελάει. Ευχαριστώ κύριε Σπρέντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τα καλά. Η απελευθέρωση των δύο συλληφθέντων μπλόγκερ ήταν θετική, αλλά πέρα από αυτό η κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν είναι πάρα πολύ αρνητική, παρενοχλούνται δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδικάζονται για ποινικά δικήματα. Μετά τις διαδηλώσεις των Πακού τον Απρίλιο έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για το Αζερβαϊτζάν γιατί το Αζερβαϊτζάν υπέγραψε τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Φαίνεται πως οι αζερικές αρχές δεν αντιλήφθησαν πως πρέπει να γίνει ένας διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να ασκεί η κυβέρνηση. Ελπίζω όμως να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με το Αζερβαϊτζάν μέσω του Euronest. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Σάκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση των δύο στο Αζερβαϊτζάν, όμως εδώ τα προβλήματα συνεχίζονται. Μα ανησυχήσαν ιδιαίτερα οι συνεχεί παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γι' αυτό οργανώσαμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Οργανώθηκαν μάλλον το Μάρτιο και τον Απρίλιο σιωπηρέ διαμαρτυρίε κατά τη κυβέρνηση. Η νεολαία, η πολιτική τη αντιπολίτευση, δημοσιογράφοι συλλαμβάνονται και κρατούνται. Ε, πολλοί διαμαρτυρητέ, ε, από του διαμαρτυρόμενου μάλλον, καταδικάστηκαν σε μαζικέ ε, δίκε και ε, πολλοί δικηγόροι δεν μπόρεσαν να μεταβούν στον τόπο εκδίκασης των υποθέσεων. Ε, δόθηκε μάλιστα διαταγή από το Υπουργείο Δικαιοσύνη να μην συνεχιστούν οι δικέ αυτέ. Αυτό το κλίμα εκφοβισμού και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να πάψει. Οι κυβερνήσεις έχουν, η κυβέρνηση μάλλον έχει καταπατήσει επανειλημμένως συμβάσει που ίδια έχει υπογράψει. Όπω ε, την ε, σύμβαση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε ο κ. Αλίγεφ να, δια... να τηρήσει τι υποσχέσει του. Διότι αλλιώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει μέτρα και θα υπάρξουν επιπτώσει στι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Αζερβαϊτζάν. Σα ευχαριστώ, Λούνα Τσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγε μέρε γιορτάσαμε στι ε, την ίδρυση του Euronest, ιδρυτικό μέλος της οποία είναι το Αζερβαϊτζάν και δεσμεύτηκε για κράτος δικαίου, ελευθερία γνώμη, συνέρχεστε τον ΜΜΕ και στο πλαίσιο της συμφωνίας ε, Σύνδεση με την Ένωση ε, αποτελεί αυτό ένα από τα βασικά της στοιχεία. Οπότε είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πώς η κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν συμπεριφέρθηκε σε ανθρώπους που διαδήλωναν ειρηνικά. Μιλάμε για νέους που οργανώθηκαν μέσω Facebook και συνελήφθησαν. Καταδικάστηκαν σε δυόμιση χρόνια φυλακή επειδή διαδήλωσαν ε, ειρηνικά υπό τον τίτλο «Χρήση ναρκωτικών» και διάφορα τέτοια. Επίσης, άλλα άτομα τα οποία διαδήλωσαν εν το μέσο της νυχτός, χωρίς δημοσιότητα και χωρίς να έχουν επαφή με δικηγόρους, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 5 μέχρι 8 χρόνια. Αυτό, κύριε Επίτροπε, είναι ανεπίτρεπτο. Ζητάμε με κοινό ψήφισμα των πέντε μεγαλύτερων ομάδων μας να αφαιθούν ελεύθερα αυτά τα άτομα, να ισχύσει το κράτος δικαίου, ελευθερία των ΜΜΕ, όπως ακριβώς ε, δεσμεύθηκε ο πρόεδρος Αλίγεφ. Και είχε πει κανένας δημοσιογράφος δεν διώκεται. Επιτέλους πρέπει να τηρηθούν αυτά και ελπίζω πώς θα επιτύχουμε μέχρι την ε, κοινοβουλευτική διάσκεψη του Ιουνίου πράγματι να φεθούν όλοι ελεύθεροι και οι συντάκτες των εφημερίδων ε, ο κύριος Φατουλάγεφ. Αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Ευχαριστούμε. Εκπρόσωπα πολιτικών ομάδων και πρώτος ο κύριος Κούκαν εκ μέρους του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση στο Αζερμπαϊτζάν πραγματικά είναι ιδιαίτερα προβληματική. Αφορά την ελευθεροτυπία, την ελευθερία έκφρασης, και πολλά άλλα προβλήματα. Έχουμε μάθει για ε, συλλήψεις, για επιθέσεις, ε, για εκφοβισμό δημοσιογράφων και άλλων ανθρώπων. Ε, το ίδιο που γίνεται και σε άλλες χώρες πρέπει να γίνει και στα Αζερμπαϊτζάν. Πρέπει να καταλάβουν εκεί ότι δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτέ οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αν η χώρα αυτή θέλει να είναι μία από τι χώρε εταίρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ε, ασπαστεί τι αξίε ε, και τι αρχέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά βέβαια φορούν την όλη περιοχή του Νότιου Καυκάσου. Θα ήθελα να σα υπενθυμίσω και την κλιμάκωση τη ένταση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία για τον Αγκόρνο Καραμπάχ που αποτελεί ένα κίνδυνο για την ασφάλεια ολόκληρη τη περιοχή εξού και ζητούμε στο ψήφισμά μα ε, να γίνουν πράγματα άμεσα και όχι μόνο στο, στην χώρα αυτή αλλά γενικότερα στην ε, περιοχή του Νότιου Καυκάσου. Θα πρέπει να δούμε και τι συνέβη ε, με τη Γεωργία. Θα πρέπει να αποφύγουμε τραγωδίες σαν αυτές που έχουν προηγηθεί. Ευχαριστώ. Βίγγενιν τώρα εκ μέρους των σοσιαλιστών. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στο Αζερβαϊτζάν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και έχουμε δίκιο να ανησυχούμε. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω την περίπτωση του κυρίου Χατζίεφ, ο οποίο ε, προσπάθησε να δώσει στι αρχέ να καταλάβουν ότι η σιωπηρή διαμαρτυρία είναι κάτι το φυσιολογικό στον πολιτικό βίο οποιασδήποτε χώρε και ότι η ποικιλία διαφορετικών πολιτικών απόψεων είναι ένα θεμελιώδη στοιχείο τη δημοκρατική κοινωνία. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι είναι λίγο ατυχέ να συζητάμε το Αζερβαϊτζάν και τη Λευκορωσία το ένα θέμα μετά το άλλο. Διότι το Αζερβαϊτζάν με τον πρόεδρο του έχει γίνει, ως, ε, έχει γίνει δεκτός ως ιδρυτής και θεμελιωτής της συνέλευσης Euronest εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν σε συνεργασία με τις αρχές ε, και την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πέραν του να ε, υιοθετούμε κατεπήγοντα ψηφίσματα. Η ευρωπαϊκή ε, συνεργασία και η πολιτική γειτονία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως κατάλληλα εργαλεία για τέτοιου είδους ε, στόχους. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέες προσδοκίες από το Αζερμπαϊτζάν, νέες ε, προσπάθειες για συζητήσει για την ειρήνη και όσα θα οργανωθούν, οι εκδηλώσει θα οργανωθούν τον Ιούνιο στο Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ω ευκαιρία για να δούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Βίγκενιν, ο κύριο Βότσον, εκ μέρου των Ελευθέρων. Κύριε Πρόεδρε, τολμώ να πω πως εάν το Αζερβαϊτζάν λεγόταν Αζερία όπως λέμε Γεωργία θα ανισχούσαν πιο πολύ οι Ευρωπαίοι. Όμως η ομάδα μου δεν συμφωνεί με την άποψη του κυρίου Βιγγένιν. Τα ΜΜΕ στο Αζερβαϊτζάν δεν είναι ελεύθερα, οι εκλογές δεν είναι δίκαιες, ε, οι άνθρωποι υπόκεινται σε αυθαιρεσίες και βία από τις αρχές. Οι ειρηνικές διαδηλώσεις τελευταίες εβδομάδες αντιμετωπίστηκαν με καταπίεση που ταιριάζει περισσότερο σε αραβική παρά σε ευρωπαϊκή χώρα. Από ένα καθεστώς 18 ετών που έχει καταπνίξει κάθε ελπίδα προόδου. Η συνεχιζόμενη συμμετοχή αυτής της χώρας στην πολιτική γειτονία πρέπει να τεθεί επιτέλους υπό τον όρο των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και όχι Τη διαθεσιμότητα πετρελαίου για τον αγωγό Ναμπούκο. Ευχαριστώ τώρα κυρία Χάουταλα για του ε, Πρασίνου. Ευχαριστώ πολύ. Η Δημοκρατία και ο σεβασμό των Ευρωπαίων δικαιωμάτων και του κράτου δικαίου είναι ένα απόσπαστο μέρο τη Νέα Συμφωνία Σύνδεση που είναι διαπραγμάτευση αυτόν τον καιρό μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν να, ε, υπάρχει χωρίς σεβασμό σε αυτές τις αρχέ, ένα κοινό μέλλον για το Αζερμπαϊτζάν και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ με του συναδέλφου που είπαν ότι πρέπει να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο και πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί όταν μιλάμε με ε, συνομιλητέ μα από τι χώρε του Νοτιού Καυκάσου να μην θεωρήσουν ότι ε, αρκεί η Λευκορωσία και κανένας άλλος δεν πρόκειται να ε, θυγεί. Η επερχόμενη μελέτη που προετοιμάζεται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, ελπίζω να μας καθοδηγήσει για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις χώρες αυτές και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το Αζερμπαϊτζάν είναι ένα ιδιαίτερο εταίρο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Euronest. Εξού και εποφελείται προνομιακών σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει λοιπόν ένα έκτακτο καθεστώς η χώρα αυτή. Όταν λοιπόν συνάπτονται μεταξύ αυτού του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνίες, θα πρέπει το κράτος αυτό να σέβεται τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, που αποτελούν προϋποθέσεις για την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξω και είναι απαράδεκτο και αδικαιολόγητο να ε, συλλαμβάνονται ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, διαδηλωτές, ε, δημοσιογράφοι ή να ασκείται βία ε, κατά των διαδηλωτών. Όπως είπε και η κυρία Άστον, μάλλον και η κυρία Άστον και η Κομισιόν πρέπει να ασκήσουν πιέση στο Αζερβαϊτζάν και πρέπει να τους μεταφέρουν τις ανησυχίες μας για την καταστολή της δημοκρατίας στη χώρα αυτή. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση ψηφίσματος Νομίζω θα πρέπει να δοθεί από την Κομισιόν η εντολή στην ΥΠΑΤ εκπρόσωπο. Ευχαριστούμε κυρία Εσάγια. Ευχαριστώ. Ε, Προεδρά και κυρία Επίτροπε, στο πλαίσιο της συνεργασίας Euronest θα πρέπει να φροντίσουμε πολύ γρήγορα να εξετάσουμε το θέμα αυτό της παραβίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θα πρέπει και στις δύο αυτές χώρες, Αζερβαϊτζάν και Λευκορωσία, να φροντίσουμε να επιβληθεί ο σεβασμός των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να υψώσουμε λίγο τους τόνους και από την άποψη των επικριτικών μας σχολείων και να έχουμε υπόψη ότι τα πράγματα εξελίσσονται και εκτός κοινοβουλίου. Μην ξεχνάτε τι συνέβη στον αραβικό κόσμο και στον αραβικό χώρο πρόσφατα. οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συνελήφθησαν, διαμαρτυρίες ε, καταπνίγηκαν και οι διαμαρτυρόμενοι πολλές φορές συνελήφθησαν. Αυτό ε, δείχνει ότι στο Αζερβαϊτζάν η κατάσταση των θεμελιωδών ελευθεριών δεν είναι σε επίπεδα ικανοποιητικά. δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. πρέπει λοιπόν να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος... Ευχαριστώ ο κύριος Κέλλη τώρα που Κύριε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. κατάσταση στο Ζερμπατζάν είναι πολύ απογοητευτική. Μιλάμε για μια χώρα που δεν έχει προοδεύσει ε, από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και είναι πολλά τα παραδείγματα ελευθερίας, ε, έλλειψης ελευθερίας του λόγου, του συνέρχεστε, ενδείξεις βασανισμού κρατουμένων, ε, δικαστικές υποθέσεις όπου χρησιμοποιούνται στοιχεία υποκλοπών, Βεβαίω, εγώ θεωρώ πέρα από το διάλογο πως όπως λέει ο κύριος Βάτσον πρέπει να φανούμε και σκληροί γιατί με αυτό το καθεστώ δεν θα πάμε πουθενά. Ναι, διάλογο αλλά πρέπει να υποβάλουμε και απαιτήσει για ελευθερία του τύπου, της έκφρασης και του συνέρχεστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Ρέπο. Ευχαριστώ πολύ. Η ελευθερία εκφρασή, η ελευθερία του συνέρχεστε αποτελούν βασικέ αρχέ, οικουμενικέ αρχέ. Το θεμέλιο ουσιαστικά τη δημοκρατία είναι οι αρχέ αυτέ και είναι κρίμα που υπάρχει παρενόχληση, απειλέ, συλλήψει και ότι όλα αυτά χρησιμοποιούνται για να ε, καταπνίξουν, ε, να ε, φημώσουν την κοινή γνώμη. Το Αζερβαϊτζάν έχει επικυρώσει την σημασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα πρέπει να σέβεται τα, τις δεσμεύσεις και τα δικαιώματα των πολιτών του. Οι blogger, οι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές, οι κοινωνία των πολιτών δεν μπορούν να εκφραστούν στη χώρα αυτή ελεύθερα, ούτε καν να διαδηλώσουν ειρηνικά μπορούν. Οι νέοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν επί παραδείγματι τις νέες τεχνολογίες επικοινωνίας ε, και τα, δίκτυα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Αζερβαϊτζάν πρέπει να σέβεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό πρέπει να είναι εγγυημένο ε, στο πλαίσιο της τελικής σχέσης μας με τη χώρα αυτή. Ο κύριος Λαντσμπέργκης είναι ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, το ψήφισμα για το Αζερβαϊτζάν εκφράζει την ανησυχία μας για πιθανές, πιθανή ηχό των γεγονότων της ε, Βορείου Αφρικής στη γειτονιά μας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με Βόρεια Αφρική, Ρωσία και Λευκορωσία θα πρέπει, μας λέτε εδώ πέρα, να αποφεύγετε. Σε ορισμένα σημεία θα μπορούσαμε να είμαστε πιο σαφείς. Οι διατυπώσεις για την κατάσταση που επιδεινώνεται ή των αυξημένο αριθμών ατυχημάτων θα πρέπει να συνοδεύονται από τη λέξη πρόσφατα. Δεν μιλάμε γενικά για το τι συμβαίνει. Αντιθέτως μέχρι τα γεγονότα αυτά τα εαρινά έκανε κάποια πρόοδο το Αζερβαϊτζάν και δεν περιελαμβανόταν από την Human Rights Watch στην κατηγορία της Κίνας, του Ιράκ, του Ισραήλ, της Ρωσίας, Σαουδικής Αραβίας, Ουσμπεκιστάν και λοιπόν το Αζερβαϊτζάν. Καλύτερα να μην αναφέρετε με αυτές τις ε, χώρες. Έτσι, λίγο πιο ισορροπημένοι να είμαστε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εγώ. Θα δώσουμε τον λόγο στην κυρία Ταντσίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Αζερβαϊτζάν είναι ένα καθοριστικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία και τη ε, συνεργασία προ Αλλά είναι και ιδρυτικό μέλο του Euronest. Θα πρέπει λοιπόν να σεβαστεί τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει έναντι τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αζερβαϊτζάν για τι θεμελιώδει ελευθερίε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου και θα πρέπει βεβαίω να μην ξεχνάμε ότι έχει υπογραφεί και η Διεθνή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ελευθερίε από το Αζερβαϊτζάν. Μιλάμε για συνθήκε τι οποίε έχει προσχωρήσει το Αζερβαϊτζάν. Μια χώρα λοιπόν η οποία θέλει να γίνει παγκοσμίω αναγνωρισμένο δημοκρατικό κράτο δεν μπορεί να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο, καταπιέζοντα και καταπνίγοντα τι διαμαρτυρίε των νέων. Δεν μπορεί να μην έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητε δίκε επειδή δεν συμφωνούν με τι ε, επικρατούσε απόψει των κυβερνώντων. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει διαρκή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει ο τύπο να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα, να αναφέρει και να ενημερώνει ξεκάθαρα και χωρίς φραγμούς την κοινή γνώμη. Θα πρέπει να ε, ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής σε αυτό το γύρο, ο κύριος Παλέτσικη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Αζερμπαϊτζάν έχει δύο πρόσωπα σήμερα. Από τη μία φαίνεται ένα, μια φαινεται αναπτυσσόμενη οικονομία με τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και πραγματικά ανοίγει για κάποιο δρόμο στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ε, Συμφωνία Σύνδεσης, ε, συμμετέχει στη συνέλευση Euronest κτλ. Από την άλλη πλευρά το άλλο πρόσωπο είναι εκφοβισμός, περιορισμός ελευθερία ε, του τύπου, συλλήψεις, όλα αυτά τα οποία ανέφεραν προλαλήσαντες. Τον Πακού θα πρέπει να ακούσει την ε, γνώμη των πολιτών του. Δεν μπορεί να είναι διπρόσωπη η χώρα και μπορεί να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τα μέσα για να το πράξει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Άντορ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι εξελίξεις. Στο Αζερβαϊτζάν όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μας ανησυχούν σοβαρά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήσαμε μία τάση αυξανόμενων περιορισμών στον τομέα αυτών. Η διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών ε, στις 7 Νοεμβρίου 2010 δεν αποτελούσε σημαντική πρόοδο στη δημοκρατική εξέλιξη της χώρας. Υπάρχουν άλλοι τομείς όπου πιστεύουμε ότι το Αζερβαϊτζάν πρέπει να βελτιώσει ε, τις προσπάθειές του για να συμμορφωθεί με τις εσμεύσεις του στον ΟΑΣΕ και Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα, ελευθερία των ΜΜΕ. Υπάρχει έλλειψη πλουραλισμού. Επίσης υπάρχουν αφορές παρενόχλησης δημοσιογράφων, και εμφυσιτούμενων ε, τακτικών. Και βεβαίω υπάρχουν και μονομένε περιπτώσει που προξενούν ανισχύ Η ελευθερία του συνέρχεστε επίση. Ένα άλλο τομέα με ανισχύει πάρα πολύ. Του τελευταίου μήνε είδαμε πάρα πολλέ σοβαρέ ε, πράξει ε, των αρχών όσον αφορά την οργανωμένη διαμαρτυρία που εμπνεύστηκαν από τις αραβικές επαναστάσεις. Η κράτηση ακτιβιστών και άλλες πράξεις καταπίεσης είναι πραγματικά λυπηρές. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ευθύνη να στείλει ένα σαφές μήνυμα για το σεβασμό της δημοκρατίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Τέτοια μηνύματα ε, ο ίδιος ο κύριος Μπαρόσο στον Πακού τον Ιανουάριο και θα είναι βεβαίως και ψηλά στις μελλοντικέ μα συζητήσεις. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι θεμέλιο της συνεργασίας μας με το Αζερβαϊτζάν σύμφωνα με την υφιστάμενη συμφωνία πέρσι. Ε, συστάθηκε μια νέα υποεπιτροπή ασφάλειας, ε, δικαιοσύνης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας και όλα αυτά αποτελούν βασικό κομμάτι των διαπραγματεύσεών μας για μια νέα συμφωνία σύνδεσης. Καλώς ορίζω την ε, διαθεσιμότητα του Αζερβαϊτζάν να συζητήσει αυτά τα ζητήματα και τον ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις δημοκρατικές αξίες ε, μέσω της ε, κοινή ε, συνεργασίας, κοινής επιτροπής συνεργασίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ κύριε Επίτροπε. Τελειώνει εδώ πέρα η συζήτηση για το Αζερβαϊτζάν. Η συζήτηση θα γίνει μετά το τέλος του επόμενου θέματος που είναι η Λευκορωσία.